Άρχεται η συνεδρίαση. Έχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο στην ε, πρώτη ανάγνωση για το θέμα του διορθωτικού προβλησμού 2019 κάθετος 08. Ε, Αυτά ε, βρίσκονται στα πρακτικά της ε, σημερινής συνεδρίασης ε, θα βρίσκονται από αύριο. Περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο των ψηφοφοριών. Έχουμε τελική ψηφοφορία για το κοινό ψήφισμα για το πι και το σχέδιο ανασυγκρότησης ψηφίζουμε τους τροπολογίες για τα εξή θέματα χρηματοδότηση των χωρών γειτονίας λόγω COVID προσωρινά μέτρα περιορισμού των αεροπορικών συγκοινωνιών ε, για την ισχύ άδειών ε, και προτύπων ε, λιμενικά τέλη, σιδηροδρομικό πακέτο. Η ψηφοφορία θα γίνει με την ίδια διαδικασία όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ο πρώτος γύρος είναι από τις 9.30 μέχρι τις 10.45. Όλες οι σημερινές ψηφοφορίες είναι ονομαστικές και τα σχετικά εγγραφά θα δημοσιευτούν σε σελίδα του Κοινοβουλίου. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 10.45 ε, και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 1 και 4. Διακόπτη συνεδρίαση.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 σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μάλιστα πολλές ε, ε, αιτήσει ε, υπευλήθησαν σε ό,τι αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή Άγκρη σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Αλίας δεν έχω δεχθεί τις ψηφοφορίες οπότε η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις Ποιος ήθελε το λόγο Έκχαρτ. Ευχαριστώ. Απλώ θα ήθελα να πω ότι ενιστάμεθα. Έχουμε αντιρρήσει ό,τι αφορά την εντολή για άμεσε διαπραγματεύσει ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια βεβαιότητα για τους γεωργούς, αλλά η Επιτροπή Άγκρη ζήτησε αντί για μονοετή διετή παράταση κάτι που προποθέτει 100 δισεκατομμύρια ευρώ διαφορά. Και η απόφαση αυτή ελήφθη στην Επιτροπή Γεωργίας. Νομίζουμε ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα που αξίζει συζήτηση στην Ολομέλεια. Δεν είμαστε κατά της ε, επέκτασης, της παράτασης, αλλά κατά της εντολής για άμεση διαπραγμάτευση, γιατί ήθελαν διαπραγμάτευση εδώ στην Ολομέλεια. Θα πίστευα. Μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει η συζήτηση να γίνει στην Ολομέλεια. Περί αυτού ψηφίζουμε. Γι' αυτό προτείνω να καταψηφίσετε το αίτημα για την εντολή, ώστε να έχουμε συζήτηση τη Ολομέλεια για το θέμα αυτό τον Ιούνιο, εγκαίρω και πολύ πριν τη λήψη τη απόφαση. Ελπίζω να με στηρίξουν στην αντίρρηση οι συνάδελφοι, να αντιληφθούν την επιχειρηματολογία και όπως είπε και ένας συνάδελφος, χρειαζόμαστε μια ισχυρή και σαφή εντολή. Και νομίζω ότι η ισχυρότερη εντολή θα δοθεί μέσω τη Ολομέλεια. Α εξασφαλίσουμε λοιπόν για τον Ιούνιο μια εντολή τη Ολομέλεια. Και γι' αυτό είμαστε κατά τη άμεση εντολή μόνο από την Επιτροπή Γεωργία για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Έκχοτ για τι διευκρινήσει. Ελπίζω να δείξετε κι εσείς μια κατανόηση γιατί κήρυξα ε, την διακοπή των εργασιών πολύ γρήγορα ε, ε, έσπευσα. Γι' αυτό βιάστηκα λίγο. Σας ζητώ συγγνώμη, ελπίζω να μην είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα το διαδικαστικό. Αυτό και τώρα πραγματικά διακόπτεται η σύνοδος.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

Il Presidente. Bonjour. Tutto bene? la galà. La seduta è ripresa. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. ιδού τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, ε, της σημερινή ψηφοφορία. Πρόταση ψηφίσματος νέο π, δελτα π, ήδη πόρη ανάκαμψη, τελική ψηφοφορία, ψηφίσαντες 693. Υπέρ 505. Κατά 119. Αποχές 69. Εγκρίνεται. μακροοικονομική βοήθεια σε χώρες ε, εταίρους ε, γειτονία και λόγω COVID-19. Τροπολογία 1 απορρίπτεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. Προσωρινά μέτρα όσον αφορά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Τροπολογία 28 απορρίπτεται. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. ένα 9, 17, 29 εγκρίνονται. 16, 22 εγκρίνονται. Τροπολογία 13, 17, 23 εγκρίνονται. Τροπολογία 29 απορρίπτεται. 4, 12, 18, 24 εγκρίνονται. Τροπολογία 5, 13, 19, 25 εγκρίνονται. 6, 14, 20, 26 εγκρίνονται. 8, 27 εγκρίνονται. Προσωρινά μέσα όσον αφορά την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών. Όμνιμπους. Τροπολογίες 4, 5, 9, 10, 11 εγκρίνονται. Τροπολογία 1, 7 απορρίπτονται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. Τροπολογία 4, 5, 6, 9, 10, 11 εγκρίνονται. Τροπολογία 2, 8 απορρίπτονται. Δικαιώματα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων. Τροπολογία 1 απορρίπτεται. Τροπολογία 16 απορρίπτεται. Τροπολογία 3, 5, 9, 11 εγκρίνονται. Τροπολογία 12 απορρίπτεται. 6, 13 απορρίπτονται. 7, 14 απορρίπτονται. Τροπολογία 17 απορρίπτεται. Τροπολογία 2, 4, 8, 10, 15 εγκρίνονται ψηφοφορία για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο παράταση των περιόδων 4, 14, 25 εγκρίνονται 5, 15, 27 εγκρίνονται 6, 16, 27 εγκρίνονται Τροπολογία 7, 17, 28 εγκρίνονται 18, 29 εγκρίνονται 8, 19, 30 εγκρίνονται. Τροπολογία 9, 20, 31 εγκρίνονται. 10, 21, 32 εγκρίνονται. 1, 11, 22 εγκρίνονται. 2, 12, 23 εγκρίνονται. 3, 13, 24 εγκρίνονται. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 14 και 15 όταν θα λάβει χώρα ο δεύτερος γύρος των ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.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 Υπότιτλοι

exists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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Η ομάδα Renew Europe διαβίβασε στον Πρόεδρο κάποιες αποφάσεις για διορισμούς σε επιτροπές θα επισυναμφθούν στα σημερινά πρακτικά και ε, τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της ανακοίνωσης τους. Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας, ε, του δεύτερου γύρου που διεξήχθη σήμερα, είναι ε, μακροοικονομική βοήθεια ε, στη γειτονία πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε μέτρα προσωρινά για υπηρεσίες εναέρειας κυκλοφορίας. Εγκρίθηκε επίση η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσωρινά μέτρα σε ό,τι αφορά ε, ε, τις άδειες και τα διπλώματα, διάφορα μέτρα. Και εδώ εγκρίθηκε η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, λιμενικά τέλη. Εγκρίθηκε επίση η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Η δέσμη μέτρων για το σιδηρόδρομο για την περίοδο εφαρμογής και εδώ εγκρίθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέλος οι μεταβατικές διατάξεις για την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, το 2021 το Ευρωπαϊκό Ταμείο συγγνώμη, για την Ανάπτυξη της Υπέθρου και το Γεωργικό Ταμείο. Η απόφαση για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις ελήφθη ε, μετά από αίτημα μιας πολιτικής ομάδας και μπορούν να αρχίσουν ε, τις διαπραγματεύσεις τους οι αρμόδιοι εξ ονόματος ε, της Επιτροπής Γεωργίας και όλου του Κοινοβουλίου. Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν χρειάζεται τρίτος γύρος ψηφοφορίας πλέον. Τα πρακτικά της συνεδρίαση 14 και 15 ε, Μαΐου θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρίαση προς έγκριση και αν δεν διαφωνείτε θα διαβιβάσω αρμοδίως τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Διακόπτεται η περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ όλες τις υπηρεσίες. Καλό σας Σαββατοκυριακό και να μείνετε όλοι υγιείς και να προσέχετε τους εαυτούς σας.